Πάμε, θα αρχίσουμε στις 3, οπότε αρχίζουμε στις 3. Λίμπε. Αγαπητοί συναδέλφοι, συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις. με την απαλλαγή των οργανισμών σε μια 8 40 της ημερήσιας διάταξης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 Λοιπόν, τώρα έχω τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Αρχίζουμε με την απαλλαγή των οργανισμών. Η συγκίτρια η Αγιάννα Ζέντερ, θέλει τον λόγο. Η συγκίτρια Ίνες, θέλεις τον λόγο. Είσαι εισηγήτρια, έτσι. Θέλεις να πάρεις το λόγο. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, όχι. Δεν ήθελα. Απλώς ε, ας περιμένουμε τρία λεπτάκια για να έρθουν οι συνάδελφοι από όλες τις μας να ψηφίσουν γιατί είναι σημαντικές ψηφορίες. Μόνο αυτό ήθελα να ζητήσω. Ε, και κάποιες άλλες μπορεί να πιο αργά. Είναι σημαντική ψηφοφορία. Ελπίζω κι εγώ, το είπα σήμερα το πρωί όμω, ότι θα αρχίσουμε στι 3, οπότε πρέπει να τηρήσουμε την ώρα, έχουμε τόσες ψηφοφορίες. Γι' αυτό, σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, οριζόντια έκθεση, λείπουν συνάδελφοι από όλε τι πολιτικές ομάδες, γι' αυτό και την τροπολογία 2 σημείο 2 της ημερήσιας διάλαξης τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές υπερψηφίστηκε υπέρ κατά αποχές τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές υπερψηφίζεται 6 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε τροπολογία 6 πρώτο μέρος έναρξη έναρξη ψηφοφορίας τροπολογία 6 πρώτο τμήμα πρώτο τμήμα τροπολογία 6 πέρα ψηφοφορίας υπερψηφίζεται Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επτά κατά απορρίφθηκε. Πού βρισκόμαστε τώρα. Τροπολογία παριθμών 8. Υπέρ. Τροπολογία 8. Έναρξη ψηφοφορίας υπέρ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 9. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει στην προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Τροπολογία παριθμών 10. είναι η οριζόντια έκθεση. Όπως είπα περισσότερες φορές, η οριζόντια έκθεση το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να σας πω πως από εδώ και πέρα θα ψηφίζετε όπως αναφέρεται στην λίστα της ψηφοφορίας. Αυτό το ονομάζουμε πειθαρχία. Παρακαλώ. Σας είπα πως θα αρχίσω τη συνεδρίαση στις 3. Έχουμε καθυστερήσει 2 λεπτά. Είναι 120 δευτερόλεπτα. Εντάξει, τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, αποδεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε 12 δεύτερο τμήμα επαλήθευση ηλεκτρονικά έναρξη πέρας της επαλήθευσης απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά Εγκρίνεται νομίζω επαλήθευση της τροπολογίας 16. 16 επαλήθευση. Η επαλήθευση έληξε. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 με προφορική τροπολογία καμία αντίρρηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 20 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως εγκρίθηκε ναι ναι ναι 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 καταπίπτει 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε 26 ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη πέρας απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνεχίζουμε με την 30 υπέρ κατά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 1, 2, υπέρ αποχές εγκρίνεται. 2, υπερκατα αποχές εγκρίνεται. 3, υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 4, υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 5, υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 6, υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. Το λιβε 1 έχει 3, υπερκατά Πρέπει να το ελέγξουμε. Λίμπε 3, έλεγχος, πρώτο τμήμα. Λίμπε 3, πρώτο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται. Το δεύτερο καλύπτεται. Λίμπε 4, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το όλο ψήφισμα, ηλεκτρονική ψήφος, έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας 20 προς 2, δύο αποχές συγχαρητήρια στον συναδελφό μας και εισηγητή, την κυρία Γιάννα Σέντα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με το 9, το σημείο 9, την Άθερ. Τροπολογία 2, απαλλαγή με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Πέρας. Και χορηγείται η απαλλαγή. Τοπολογία ε, 3 και 4 καταπίπτουν. Και τώρα για την απόφαση απαλλαγής άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Χορηγείται με την ίδια πλειοψηφία. Και για το κλείσιμο των λογαριασμών δεν απαιτείται ψηφοφορία. Δηλαδή εξυπονοείται. Λοιπόν, σε τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχε... αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές δεν κρυπτεί. Τροπολογία 18, καταπίπτει. 19 υπέρ, κατά. Α, δεν καταπίπτει, συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε την 18. Συγγνώμη. 18. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές.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 αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται 19 με 5. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ε, Μπερέκ. Ε, Φορέα ε, ρυθμιστών. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την απόφαση απαλλαγή στο σύνολό τη με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. μας λείπει κάποιος ακόμα, ένα άτομο. Πατήστε το κουμπάκι. Πέρασε. 19 υπέρ 5 κατά, ευχαριστώ. Άρα, υπονοείται το κλείσιμο των λογαριασμών. Ξεκινάμε ψήφισμα 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ όχι 13 συγγνώμη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ Όχι, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. 20 υπέρ 3 Κατά συγχαρητήρια. Το μεταφραστικό κέντρο. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την απαλλαγή στο σύνολό της με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Απόφαση για να κλείσουν λογαριασμοί εννοείται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τα 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 21 με 3, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σεντεφόπ. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την απόφαση απαλλαγή. Πέρα 21 με 4. Ωραία. Άρα κλείνουν και οι λογαριασμοί. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 7 υπέρ Κατά. Πρέπει να την επαληθέσουμε η Τροπολογία 7. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 1 καλύπτεται, έμπλ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 5 καλύπτεται. Έμπλ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 8 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Έμπλ 9 καλύπτεται. Ψηφίζουμε το ψήσιμο σύνολό του. Μονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. 22 υπέρ, 3 κατά, συγχαρητήρια, Σέπολ. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απαλλαγή στο σύνολό της μενομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. 22 με 4. Άρα κλείνουν και οι λογαριασμοί. Ψήφισμα, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά πρέπει να επαληθεύσουμε 10 νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά δεν είμαι σίγουρη Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 1 και Λίμπε 2 καλύπτονται. Λίμπε 3 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεν υπάρχει δεύτερο μέρος. Τροπολογία. Λίμπε 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 6 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την Λίμπε 6. Πέρας. Ε, είχε περάσει. Εάζα. Τροπολογία 1 υπέρ. Α, ναι. Όχι, συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Mm. Πέρας. 22, 5 κατά. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ που προσέχετε. Εάζα. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή απαλλαγή με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας 22.05 ευχαριστώ πάρα πολύ κλείνουν και οι λογαριασμοί ψήφισμα τοπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 ε, καταπίπτει. 13 σε 2 μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 και 19 αποσύρονται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 1 έως 3 καλύπτονται τραν 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τραν 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τραν 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τραν 7 ε, υπέρ, κατά αποχές 11 και 12 καλύπτονται, το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, είμαι έτοιμη να σας ζητήσω μπλοκ, αλλά ξέρω ότι μετά θα υπάρχει πρόβλημα. Don't hesitate speed up. Γρήγορα, γρήγορα. Ε, μετράει ακόμα το μηχάνημα, δεν, δεν ξέρω τι γίνεται. Πατήστε το κουμπάκι παρακαλώ όλοι. Είμαστε 27. Εδώ εσείς κολλησιεργείτε. Λοιπόν, 22 με 4. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εάζω. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεν Απαλλαγή με νομαστική ψηφοφορία άρχεται. Θα με γκρουμονείτε, λέει, χρόνο γλιτώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγκρίνεται. Κλείνουν και οι λογαριασμοί. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αυτή πρέπει να τη ξαναδούμε λοιπόν τροπολογία 12 Πέρας. Απορρίφθηκε. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 16 καταπίπτει. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 19 καταπίπτει. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 1 και 2 καλύπτονται, Λίμπε 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Λίμπε 4 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 6 καλύπτει. Λίμπε 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Στον συγητή Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο καταπίπτει. Ε, Λεωπόφαση απαλλαγής με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχιτή ψηφοφορία. Κλείνουν και οι λογαριασμοί. τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Την 9. Και πέρα και εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πέρασε αλλά να το επαληθεύσουμε 12 Πέρας, απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 καταπλήκτη 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές ποιος ήταν υπέρ 23 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίθηκε. 24. Ναι. Λοιπόν, να επαληθεύσουμε την 23. 13 υπέρ 11 κατά. Μα αργεί το μηχάνημα. Λοιπόν, εγκρίθηκε. Η 23 ήταν αυτή, ε? ναι. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απολύπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απολύπτεται. Η 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκον 1 υπέρ αποχές, ε, ε, έκον 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκον 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκον 4 καταπίπτει έκον 5 έως 7 μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 8 ε, και 9 καταπίπτουν, έχουν 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήσιμο σύνολό του μονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πατήσατε όλο το κουμπάκι. Ωραία. Ναι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον συγητή. Η CDC. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απαλλαγή με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Απολογία. Τρία. Ε, 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 είπε σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. NV1 και 2 καλύπτονται. Μπορούμε να κάνουμε μπλοκ 3-12. Ε, έως 11, όλες μαζί. Ναι, ωραία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται το ψήφισμα στο σύνολό του μονασχή ψηφοφορία άρχεται Πέρασε. 23 με 4, συγχαρητήρια, ΕΚΑ. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα με τροπολογία 18. Ο εισηγητής δεν συμφωνεί με την κλασική τροποποίηση που είχε κατατεθεί. Ε, και άρα ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Τροπολογία 18. Το έχετε στον κατάλογο ψηφοφοριών. που λέει αναγνωρίζει το ότι η ισορροπία των φύλων στα ΔΣ του υπηρεσία είναι 44 56%. Ψηφίζουμε λοιπόν την αρχική τροπολογία. Δεν έγινε δεκτή η γλωσσική εκδοχή από τον εισηγητή. Ναι. Δεν πρέπει να παίρνουν καλά οι διερμηνείς. Λοιπόν. Πάντα υπάρχει μία έκπληξη. Λοιπόν, τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δύο Καταπίπτει. Ονομαστική ψηφοφορία. Η απόφαση απαλλαγής. Πέρας. 21 με 5, ευχαριστώ. Κλείνουν και οι λογαριασμοί. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8 αποσύρεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Καμία αντίρρηση όχι. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 και 11 αποσύρονται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 18 πέρας και απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε με την ίδια πλειοψηφία να την επαληθεύσουμε 19 Πέρας. Εγκρίθηκε. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV1 έως 5. Να το κάνουμε όλα μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. NV6 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV7 μέχρι 13 η 9 καλύπτεται. Να τις κάνουμε μπλοκ. Όλες μαζί. 7 με 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 καλύπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα είστε πιο γρήγορα από μένα 22 με 5 συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται για την υπηρεσία περιβάλλοντο, Απαλλαγή με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρα. 21 6. Το κλείσιμο των λογαριασμών. Λοιπόν, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχέ απορρίφθηκε. 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Να δούμε το 12. Απορρίπτεται νομίζω. 12. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 14 και 15 αποσύρονται, συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, ναι, ναι. 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ, κατά αποχές 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. NV1 καλύπτεται. NV2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. NV3 καλύπτεται. NV4 με 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. NV7 καλύπτεται. NV8 έως 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Και κάνουμε το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε. 23, με 4, συγχαρητήρια. Εύκα. Ε, υπηρεσία αλληλεία. Σπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Απόφαση απαλλαγή με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. Πέρασε ψηφοφορία. Έχετε η απαλλαγή. Κλείσιμο λογαριασμών. Τροπολογία 6 υπέρ κατά ε, ε, ε, εγκρίνεται 7 εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πες ενευτρία καλύπτεται 4 υπέρ κατά έλεγχος για την αλίας υπαριθμών 4 νομίζω απορρίπτεται έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Πες 5 καλύτερα. Πες έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να κάνουμε έλεγχο. Πες έξι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πες επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 9 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πες 9 πέρας εγκρίνεται. Πες 10 καλύπτεται και 11. Πες 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Το πες 15. Μια φορά μετά το 12 την πλειοψηφία. Ε, απορρίπτεται. 16 καλύπτεται. Το σύντομο ψήφισμα είναι το σωμαστική. Ψηφίζουμε. σου. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Εύσα. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η απόφαση της απαλλαγής, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Χορηγείται και κλείσιμο λογαριασμό. Το πρώτο του ψηφίσματος. Εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 ε, υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά. Έλεγχος. Για το 13. 13. Έλεγχος. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ε, εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 25. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Προηγούμενο. 24. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Η 26 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Έλεγχος για το 26. Δεν μπορώ να διακρίνω, δεν ξέρω αν ε, εγκρίθηκε. Όχι, ναι, ναι, εγκρίθηκε όντως. 27. Υπέρ, κατά, αποχές. Α, 28. Υπέρ, κατά, αποχές. Α, απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά άποχέ απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά άποχέ απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά. Έρχομαι το 38, νομίζω είναι.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 εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά άποχε. απορρίπτεται. 8 υπέρ Αποχέ. αποχές Ενβι NV4, 5 και 6 μαζί. 4, 5, 6. Όλε μαζι μαζί υπέρ Αποχέ. αποχές Ενβι 7 NV7 υπέρ Αποχέ. αποχές Ενβι NV8 υπέρ Αποχέ. αποχές Ενβι NV9 υπέρ Αποχέ. αποχές Ενβι NV10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 με 15 Δεσέμβρη όλες μαζί το 12 χωριστά το 11 το 12 ε, το 11, το 11, συγγνώμη. Ε, το 11 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρινεται Ενβι NV13 υπέρ κατά αποχές Ενβι NV14 υπέρ κατά αποχές Ενβι NV15 υπέρ κατά αποχές Ενβι NV16 καλύπτεται το σύνολο του ψηφίσματος όρο στη ψηφορία. Πέρας. 23-5. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Άγγια. Ισότητα φίλων. Υπέρ κατά... Ε, τώρα και τώρα η απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής. Υπέρ. Κατά. Πέρας. Ευχαριστώ. μας κλείνουν οι λογαριασμοί. Τροπολογία 6, κατά. Τροπολογία 7 εγκρίνεται προηγούμενη, απορρίπτεται η 7, η 8 τώρα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 10 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται, 11 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 12 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 14 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Φαμ ένα καλύπτεται, 2 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Φαμ 3 και τέσσερα καλύπτεται. φαμ 5 μέχρι 9. Όλες μαζί, μάλιστα. Φαμ 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Φαμ 6 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. Φαμ 7 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. Φαμ 8 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται εγκρίνεται φαμ 9 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φαμ 10 καλύπτονται το ψήφισμα με νοστική ψηφοφορία πέρασε 23 συγχαρητήρια στον συγκεκριτή και τώρα ΑΙΟΠΑ ασφάλιες τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Απόφαση απαλλαγή ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. περασε 22-5. Ευχαριστώ. Κλείσιμο λογαριασμών επομένω. Το ψήφισμα. 6 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 καταπέπτει 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά 20 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 2 με έκον 9 μαζί μάλιστα. Ένα με έξι. Προτείνει Μαριά. υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Έχουν 7 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Έχουν 8 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Έχουν 9 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματο με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Γιατί. Ένα υπέρ κατά αποχές από ονομαστική ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται κλεισμό 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 σε δύο τμήματα Πρώτο υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρκατα αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ αποχές απορρίπτεται. 12 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Το 13 κατά το 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Έξι ε, έξι εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συναντήρια στην συγκέντρια. Ήμα. Πεθμονέων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απόφαση απαλλαγή, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρα Εγκρίνεται. Κλείσιμο βιασμών. Τροπολογία 6 υπερκατα Α, απορρίπτεται. 7 υπερθέτα αποχέ Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά ε, Απορρίπτεται. 9 υπερκατα κατά Απορρίπτεται. 9 10, 10. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 14. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16. Υπέρ κατά άποχέ. απορρίπτεται. 17. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 αποσύρθηκε. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω εγκρίνεται. Έλεγχος. Για το 22. Check is over. It is adopted, sorry. Amendment... Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV2 καλύπτεται. NV3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 καλύπτεται. 5 της NV εγκρίνεται. NV6 καλύπτεται. Θέλετε NV7 με 10 μαζί. 7 με 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. NV11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV 14 καλύπτε το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία. And it is 23 to 5. 23-5 συγχαρητήρια συγκεντρία. Κέντρο Παγκόσμιου Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απόφαση απαλλαγής. Είμαστε ψηφοφορία Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται την τροπολογία υπέρ, εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 1 με 5 καλύπτονται λίμπε 6 με 8 μαζί όχι λίμπε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 της λίμπε καλύπτεται το ψήφισμα νομαστική ψηφοφορία 24 4. Congratulations to the 24 4 στην συγκήτρια. Έμσα. Ένα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η απαλλαγή. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφορίας εγκρίνεται οπότε και το κλείσιμο των λογαριασμών τροπολογία 6 υπερκατά εγκρίθηκε συμβαστική 1 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 9 καταπίπτει 10 σε δύο μέρη πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπερκατά απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά επαλήθευση τροπολογία 12 ας την επαληθεύσουμε πέρας εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 1 έως τραν 5 καλύπτονται τραν 6 έως τραν 8 μαζί ναι τραν 6 έως 8 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 39 έως 10 καλύπτονται η όλοι το όλο ψήφισμα μεσονομαστικής ψηφοφορίας πέρας 24 προς 4 συγχαρητήρια στον εισηγητή ενίσα τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απόφαση απαλλαγής μεσονομαστικής ψηφοφορίας Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται, περιλαμβάνει το χρήσιμο των λογαριασμών, τροπολογία 6 υπέρ κατά εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 καταπίπτει, 14 δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπερκατά αποχές απορρίπτεται 15 υπερκατά αποχές απορρίπτεται 16 υπερ κατά αποχές εγκρίνεται 17 16 καταπίπτει, 17 υπερκατά εγκρίνεται, 5 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Όλο το ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη. Λείπει ένας ακόμα. Πέρας. Συγχαρητήρια στον εισηγήτη. Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τροπολογία 1 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα απαλλαγής έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται περιλαμβάνει το κλείσιμο των λογαριασμών τροπολογία 6 υπέρ κατά νομίζω απορρίφθηκε να το επαληθεύσουμε την τροπολογία 6 πέρας επαλήθευσης απορρίπτεται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 13 επαλήθευση. Πέρας επαλήθευσης εγκρίνεται. για 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 1 και 2 καλύπτονται τραν 3 και 4 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 πέρας εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευρατών, τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η απόφαση απαλλαγής με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη, πέρας. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει το κλείσιμο των λογαριασμών. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε επί του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έσμα τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ψηφίζουμε επί της απόφασης απαλλαγής μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας έναρξη πέρας εγκρίνεται το οποίο σημαίνει και το κλείσιμο των λογαριασμών τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ 8 αποχές ε, εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ναι, τροπολογία 10 επαλήθευση. Πέρας επαλήθευσης με πλειοψηφία μιας ψήφου απορρίπτεται, συγγνώμη, συμβιβαστική 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 καταπίπτει, 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έκον 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έκον 2 καλύπτεται, έκον 3 έως έκον 8 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη, πέρας, 25 προς 4, ETF. Ε Ένα υπερκατά αποχές εγκρίνεται, αποφασία απαλλαγής, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη, Το μηχάνημα ακόμα δεν έχει μετρήσει δύο. Πέρας. Πέρας ψηφοφορίας, ναι. 23 προς 4. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσιμο λογαριασμών έγινε. Ψήφισμα τροπολογία 7 υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπερ... Καταπίπτει μάλλον. 11 καταπίπτει, 12 υπέρ, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλε ανακαλύπτεται, έμπλε 2 έως 6, όλα μαζί, εν μπλοκ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 και 8 καλύπτονται, ονομαστική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος, έναρξη. Πέρας εγκρίνεται με μεγάλη ψηφοφορία συγχαρητήρια. Η Γιουλίζα, τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αποφάση απαλλαγής με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. 20. Εγκρίνεται σημαίνει κλείσιμο λογαριασμών. Τροπολογία 6 με προφορική τροπολογία αντιρρήσεις όχι υπέρ... Ναι. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Τροπολογία 6 με προφορική τροπολογία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ εν, κατά αποχές επαλήθευση τροπολογίας 8. Μπορούμε να την επαληθεύσουμε. απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 καταπίτη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 1 έως 3 καλύπτονται, Λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Λίμπε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Λίμπε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το ψηφίσμα μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας, έναρξη, πέρας, 25 προς 4, καλή πλειοψηφία, συγχαρητήρια στον εισηγητή. EU όσα, τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απόφαση απαλλαγής, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη, πέρας, 25 προς 4 έγινε το κλείσιμο των λογαριασμών τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 καταπίπτει 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 1 πρώτο μέρος θα ψηφίσουμε για το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλ 3 5 καλύπτονται, έμπλ 6 εγκρίνεται. Το ψήφισμα μέσω μαζικής ψηφοφορίας άρχεται. Ναι, είναι ένας περισσότερος από το SND. πέρας 25 προς 4 συγχαρητήρια στον εισηγητή Eurofound τροπολογία 1 εγκρίνεται απόφαση απαλλαγής μεσονομαστικής ψηφοφορίας έναρξη πέρας εγκρίνεται, γίνεται το κλείσιμο λογαριασμών, 1 εγκρίνεται, τροπολογία 9, τροπολογία 12, εγκρίνεται 13, ε, αποσύρθηκε 14 υπέρ κατά εγκρίνεται, 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 16 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το επαληθεύσουμε την τροπολογία 16, επαλήθευση τροπολογίας 16 ναι, πέρας επαλήθευση. απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές. 17 υπέρ, κατά. Ναι. 17 πρέπει να την επαληθεύσουμε, συγγνώμη. Τροπολογία 17. Επαλήθευση.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 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλ 1 καλύπτεται, έμπλ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλ 4 σε 7 καλύπτονται, το ψήφισμα μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας η οποία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Eurojust. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απόφαση απαλλαγή, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία, κλείσιμο των λογαριασμών έγινε, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ πρέπει να το επαληθεύσουμε την 11 επαλήθευση πέρας επαλήθευσης εγκρίνεται όχι απορρίπτεται συγγνώμη απορρίπτεται Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 1 καλύπτεται. Λίμπε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 5 καλύπτεται. Λίμπε 6 υπέρ κατά αποχές Λίμπε 6 θέμου, αυτό είναι να περιθέψουμε. πέρας απαλήθευσης εγκρίνεται. Το ψηφίσμα μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας άρχεται πέρας πέρας ψηφοφορίας με ευρία πλειοψηφία εγκρίνεται συγχαρητήρια. Ευρωπόλ, τροπολογία 1 επερκατά κατά αποχές εγκρίνεται, η απόφαση απαλλαγής μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει κλείσιμο λογαριασμών. Ε, τροπολογία 6 υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 6, 7 υπερκατά εγκρίνεται, 8 υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπερκατά αποχές ε, απορρίπτεται, 5 υπερκατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 1 και 2 καλύπτονται, λίμπε 3 Πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 4 υπέρ. Νομίζω απορρίπτεται. Λίμπε 5 επαλήθευση. Πέρασε επαλήθευσης. Εγκρίνεται. Λίβε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Λίβε 8 υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται, Λίβε 9 υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται. Και το ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη, πέρας, 25 προς 4, συγχαρητήρια. Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τροπολογία 1 υπερκατά αποχές εγκρίνεται, αποφασία απαλλαγής,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 κατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, λίμπε 8 καλύπτεται, λίμπε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας, έναρξη πέρας εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Frontex, τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η απόφαση απαλλαγής με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη. Λείπει κάποιος. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται, το οποίο σημαίνει κλείσιμο λογαριασμών. Ψήφισμα το 5 εγκρίθηκε, 6 υπερκατά εγκρίθηκε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ με προφορική τροπολογία χωρίς αντιρρήσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 Πληροφορία κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπερκατά εγκρίνεται, δεύτερο υπερκατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ναι 13 ναι πέρας επαλήθευσης εγκρίνεται λίμπε 1 έως 3 καλύπτονται λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 5 υπέρ λίμπε 7 συγγνώμη 7 εγκρίθηκε λίμπε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λίμπε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα συνολικά μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας η οποία άρχεται πέρας ψηφοφορίας μεγάλη φιλοψηφία έγκριση συγχαρητήρια στον εισηγητή GNSS ναι, καταπίπτει. Ναι, συγγνώμη, καταπίπτει. GNSS. Τροπολογία να υπερκάτα κατά αποχές εγκρίνεται. Απόφαση μέσω ορματική ψηφοφορία, η οποία άρχεται. Πέρας. Αυτό σημαίνει κλείσιμο λογαριασμών.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 εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 καταπίπτει 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 καταπίπτει 20 καταπίπτει Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το όλο ψήφισμα μέσω μαστικής ψηφοφορίας άρχεται πέρας συγχαρητήρια στον εισηγητή κύριε Μάτιας παρακαλώ στην uh, I will speak yeah. uh, <laughs> κυρία Πρόεδρε στην uh, ψηφοφορία που έχουμε για το draft report για το budget της ε, Parliament, Section 1 Parliament, European Parliament, ε, στην ε, τροπολογία 3 δεν έχει αναφέρει η γραμματεία κατά λάθο το όνομά μου. Αναφέρει τους συναδέλφους Σαρνιέσκι Φίτο, Σούλικ, Γκοσγεύκα, και επίσης πρέπει να προσθέσει και το όνομά μου. Έχω καταθέσει και εγώ την τροπολογία αυτή. Okay. You talk about Amendment 3. I'm talking about Amendment 3. Yeah. The, the, the Secretariat has to, to add yeah. my name. Ναι, ε, πρέπει να προσθέσει η γραμματεία το όνομά μου. Ναι, την υπέγραψα, ναι, βεβαίω. Οκ, okay, εντάξει. Βεβαίω θα το διορθώσουμε. Λοιπόν, έχετε τους καταλόγους ε, ψηφοφορίας. Συνεχίζουμε με την απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Η συγητής είναι ο κ. Δεγιόγκ. Θέλει το λόγο. Όχι, ξεκινάμε λοιπόν. Amendment, Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, απόφαση απαλλαγής ε, με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λείπουν δύο ακόμα. Πέρας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος λείπει. 27. Κάποιος άλλος, όχι. Πέρασε. Δεν λοιπόν η επιλογή. Το ψήφισμα. Αυτό σημαίνει βεβαίως... Ναι, τώρα απολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, να το κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχέ συγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχέ συγκρίνεται. 8 και 9 μαζί υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτονται. 10 καταπίπτει. 11 καταπίπτει. 12 αποσύρεται. 13 υπέρ. Κατά Να την επαληθεύσουμε. Ναι, δεν είναι σαφές ποιος είναι υπέρ. Μάλιστα. Πέρασε. Εγκρίνεται. 14 καταπίπτει, 16. Χωριστή ψηφοφορία, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ, κατά εποχέ εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 17 κατά πίπτη 18 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά. 18 Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. 18 κατά απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20. Να Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 καταπίπτει. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 καταπίπτει. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται σε δύο μέρη. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές. Ναι, ναι. Να την επαληθεύσουμε. 28. Την επαληθεύουμε. πέρας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 39. Εγκρίνεται. 40 καταπίπτει. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι, ναι. Να την επαληθεύσουμε. 42. 42 την επαληθεύουμε. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, συγγνώμη. 43 επέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 44 πέρ, κατά. Να το επαληθεύσουμε, νομίζω ότι εγκρίνεται. 44. Εγκρίνεται. 45 καταπίπτει, 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 47 την επαληθεύουμε ηλεκτρονικά εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52. Να, να επαληθεύσουμε την 50. 50. Πέρας. Απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51, να την επαληθεύσουμε. Πέρας, 17 υπέρ. 53 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, ναι. Να την επαληθεύσουμε 53. ...54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ναι ναι πάει 54 να την επαληθεύσουμε πέρας εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε την 55 55 ναι. πέρας εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 αποσύρεται 57 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 αποσύρεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι. 61. Επαλήθευση. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 κατά αποχές. Λοιπόν, συμβαστική δύο να τα παληθεύσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, συμβαστική ε, τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68, 69, 70 κτλ 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 καταπίπτει Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά αποχές ε, γκρίνεται, Ο 86 σε δύο μέρη. μέρο πρώτο. Υπέρ. Κατά αποχέ. Να το επαληθεύσουμε το 86. Μέρος πρώτο. εγκρίνεται. Μέρο ε, δεύτερον προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά 87 υπέρ, κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 91 έω 95 Κατά. Ε, Ζήτησαμε ονομαστική ψηφοφορία για την 91 έως 95. Είχε υποβληθεί στην γραμματεία με τους συναδέλφους Τάς, Ντεγιόγκ, Φλάναγκαν, Πετιτσίνη και ε, πρέπει να, ναι, ναι, υπάρχουν έξι βουλευτές που στηρίζουν το αίτημα. Ποιοι είναι. Μάλιστα. Ωραία. Ονομαστική ψηφοφορία. 91 έως 95 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτονται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90 91 έως 95 απορρίφθηκαν. Γι' αυτό περάσαμε στην 89. Η 89 εγκρίθηκε. Να το επαληθεύσω αν έχετε αμφιβολία. Τροπολογία 90. Καταπίπτει. Και τώρα έχουμε τροπολογία 96, 97. Καταπίπτει. 97. 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 καταπίπτει. 99 καταπίπτει. 100 καταπίπτει. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 καταπίπτει. 103 καταπίπτει. 104 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Για ναι, να το ξαναδούμε. 104, ναι. Πέρας, απορρίπτονται. 105 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά πίπτη 110 υπέρ κατά αποχές 111 και 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ 114 υπέρ μέχρι 17 ε, αποσύρονται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120, 121 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, ορίστε. Ναι, να την επαληθεύσουμε. 122 λοιπόν. Πέρας. Απορρίπτεται. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 127 κατά καταπίπτει. Και συνεχίζουμε με τη συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την 100. Τι είπατε? Πώς? 147 υπέρ. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 και 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 και 152 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 151 και το 152 Πέρας εγκρίνεται 153 και 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την πλειοψηφία 155 κατά πίπτη 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Έλεγχος για το 158. πέρας Απορρίπτεται. 160 και 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Έλεγχος. Έχει κανείς να το εκτιμηθεί του ως πρόεδρος, την περηφάνεια του. It is rejected. Απορρίπτωση. 159. Υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγχος. Δεν μπορώ να διακρίνω. 159. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 163 163. Εγκρίνεται. Με ένα ψήφο, μία ψήφο τέλο πάντων, 164. Καταπίπτει 165. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 166. Αποσύρεται. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι 68 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 169. Καταπίπτει. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, κα, πώς? Μάλιστα. 170. 170. Έλεγχος. Πέρας. Είναι 171 υπέρ. Κατά. αποχές. Εγκρίνεται. 172 και 173 καταπίπτουν. 174 υπέρ. Κατά. αποχές. απολύτως. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Νομίζω. 175. Πέρας. Απορρίπτεται. 176. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178. Υπέρ. Κατά. Αποχές για το 178. Απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για το 180. Έλεγχος. Πέρας εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. 182. Απορρίπτεται. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ζωτέ απορρίπτεται, αλλά ας ε, ελέγξουμε 183. Εγκρίνεται. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 το διάφορο και πάμε στο 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι αποσύρεται έλεγχος 194 έλεγχος 194 επαναλαμβάνει η πρόεδρος πέρας εγκρίνεται 195 εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Απορρίπτω η επόμενη 199 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 199. 200 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Νομίζω εγκρίνεται έλεγχος. Έλεγχος για το 200. Εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 έλεγχος. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. 23 καταπίπτει, 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές αν εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος 208 208 πέρασε εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 209. Πέρασε. και σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 κατά πίπτη 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 218 πίπτη, 219 ε, εγκρίνεται. 220-221 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 221 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 223 καταπίπτει. 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 έλεγχος. Εγκρίνεται, ναι. 228 υπέρ κατά έλεγχος για το 228 228 Εγκρίνεται. 229 εγκρίνεται υπέρ κατά εγκρίνεται το 31 υπέρ κατά εγκρίνεται ναι, ναι, 231 έλεγχος έλεγχος πέρας και «232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 233 το δύο τμήματα. Το πρώτο. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Περ κατά αποχές εγκρίνεται. 234 κατά πίπτη, 235 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 236 σε τμήματα, το πρώτο υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, του 236. Δεύτερο τμήμα του 236. Ε, Πέρας του ελέγχου. Και απορρίπτεται. 237 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 238 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 239 έλεγχος Δεν ξέρω ποιος κέρδισε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Νομίζω πάντως ότι εγκρίνεται. Ναι, έτσι είναι. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 240. Έλεγχος. Ναι, εγκρίνεται. 241. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 242. 242 έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά 242. It is adopted. 243 in favor, against. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 244, υπέρ, κατά, αποχές. 244. It is adopted. 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό 246 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται για να δούμε 246 δεν προβλεπόταν. Ποιος είναι τα αυτό; Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 241 καταβλήτη, 250. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 251 in favor. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 252 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 253 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.55 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 2.55 έλεγχος Πέρασε απορρίπτεται 2.56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.57 και 2.58 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Α, όχι, όχι, λάθος. Κατά πίπτη. 2.59 υπέρ. Εγκρίνεται. 2.60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,66 καταπίπτει. 2,67 έως 2,60 από κοινού. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 2,71 καταπίπτει. 2,72 επίση. 1 υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματο. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζομαι. Open. The vote is open. The vote is closed. Πέρασε. Congratulations to the rapporteur. Thank you very much. Now what we do... Και σας ευχαριστώ. Yeah, now we vote, now we vote on the external action service. Για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχετε λάβει τους καταλόγους για την ψηφορία. Other institutions. Ah ja, alles klar. Ja, okay. Ich habe gefragt. Ja, okay. We vote. Ja. Ja. Das ist mit Ihnen Genau. Ja. We vote now other institutions. If you continue with a little bit of discipline, we will have, we'll be able to escape soon. Θα τελειώσουμε σύντομα, εάν επιδείξετε επιθαρχία. Other institutions. Άλλα θεσμικά όργανα. Other institutions. The rapporteurs Bart Stas and Benedict Yavo. Do the rapporteurs wish to take the floor? Θέλουν να λάβουν το λόγο. Άλλα θεσμικά όργανα, εισηγητέ. Ωραία, πάμε τότε στην υπηρεσία εξωτερική δράση και ψηφίσουμε για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επομένως. Πάμε κατευθείαν στην απόφαση της απαλλαγής. Όχι, όχι. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η απόφαση της απαλλαγής. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. We vote on this, yeah, discharge by roll call. Παλαίμενο στην ψηφοφορία. Λοιπόν. λοιπόν, δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Still two members missing. Ακόμη δεν έχουν ψηφίσει αυτοί οι δύο συνάδελφοι. It would be great to, to draw out the cards really. Okay, the vote is closed. Πέρασε. 20 to 4, thank you.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 233 3 Συγχαρητήρια. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και Συμβούλιο. Το συν σημαίνει αναβολή. Δεν έχουμε τροπολογίες και πάμε ευθύς στην ψηφορία για την απαλλαγή. Ψηφίζουμε. Το συν σημαίνει αναβολή. Είπαμε. Το πλήν σημαίνει χορήγηση της απαλλαγής. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. If you, yeah. If you vote, if you vote, yeah. Yeah. Yeah. If you, if you vote, if you vote minus, you... Να ψηφίσετε κατά σημαίνει ότι χορηγείτε την απαλλαγή αν ψηφίσετε υπέρ, αναβάλλετε τη χορηγή τη απαλλαγή. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. If you want to postpone, you need to change your vote. Yeah. Yeah. Anything else unclear? Ποιος δεν καταλαβαίνει κάτι. Λείπουν δύο συνάδελφοι ακόμη. Uh, manchmal. Okay. The vote is closed. Πέρα ψηφορίες. Αυτό είναι σωστή αφετηρία για διαπραγματεύσει. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορια Ψηφίζουμε. The vote περα ψηφοφορία. ψηφορίες. Τώρα, τώρα. 22-1. Συγχαρητήρια. Justice. Yeah. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. μόνο δύο τροπολογία. Υπέρ. Κατά. αποχή. Εγκρίνεται. Απόφαση χορήγησης της απαλλαγής, ομοιονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ένα, υπέρ, κατά. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Αποσύρεται. Ε, πέντε εγκρίνεται, έξι υπέρ κατά. Αποχές Έλεγχος για το 6. And it is adopted. Amendment 7. Το 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 9.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 16. Υπέρ κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 16. 16. Πέρασε. Απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Νομίζω απορρίπτεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 καταπίπτει. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος μειονομαστική ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ελεγκτικό συνέδριο Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 και 3 καταπίπτουν. Απόφαση απαλλαγής μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας. The vote is closed. And it is granted. Εγκρίνεται το ψήφισμα τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ 8 αποχές να το ελέγξουμε τροπολογία 7 τροπολογία 7 τροπολογία 7 ας το ελέγξουμε Πέρας επαλήθευσης εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 10 σε 4 μέρη. Πρώτο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τρίτο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τέταρτο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 με προφορική τροπολογία χωρίς αντιρρήσεις υπέρ κατά ο τροπολογία 12 επαλήθευση νομίζω πως εγκρίθηκε αλλά ναι πέρασε επαλήθευση, ναι εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά Ας το επαληθεύσουμε. 15. Ας επαληθεύσουμε την 15. Ναι. Πέρας επαλήθευσης εγκρίνεται, συγγνώμη.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 25 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται ας επαληθεύσουμε μπορούμε να επαληθεύσουμε ξανά την 25 πέρας επαλήθευσης ναι εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά νομίζω πως εγκρίθηκε αλλά θα πρέπει να την επαληθεύσουμε 27. Τροπολογία 27. Τροπολογία 27. Πέρασε παρήθεση, εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επί του συνόλου του ψηφίσματος μεσονομαστικής ψηφοφορίας Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται απόφαση απαλλαγη με ψηφοφορία άρχεται πέρας 22 προς 4 ευχαριστώ το ψήφισμα τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ναι, θα ελέγξουμε την τροπολογία 5. Την ελέγχουμε. πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά Ας επαληθεύσουμε την τροπολογία 9. Ας την επαληθεύσουμε την 9. Πέρας. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 12. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε την τροπολογία 12. πατέρας Εγκρίνεται, με ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. 13 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας άρχεται. 23 από 3, συγχαρητήρια στους εισηγητές. Επιτροπή των Περιφερειών, τροπολογία 1 και 2, υπερκατά κατά αποχές απορρίπτεται. Απόφαση απαλλαγής μεσονομαστικής ψηφοφορίας άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Το ψήφισμα, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ 9 8 κατά εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ ναι ναι να επαληθεύσουμε την τροπολογία 10 πέρας εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 κατά πίπτη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας άρχεται πέρας 23 προς 3 συγχαρητήρια στον διαμεσοβαλή ο διαμεσολαβητής ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται ονομαστική ψηφοφορία η απόψη επαλλαγής άρχεται 25 προς 1. Πέρασε. Ευχαριστώ. Το ψήφισμα. υπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να την επαληθεύσουμε. Επαληθεύσουμε την 5. 5. Ευχαριστώ, απορρίπτεται, συγγνώμη. Δεν ήταν σαφές. Γιατί δεν βλέπω όλη την... όλα τα χέρια. Έξι υπέρ. Κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική σοφορία. άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Επόπτης προσωπικών δεδομένων τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η απόφαση απαλλαγής με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας ευχαριστώ ψήφισμα τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ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 Μπορούμε να τα ψήσουμε όλα μαζί. Έξι υπέρ κατά... Εφτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 έως 12 μαζί, όλες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια στους συζητητές. Μπορούμε να κάνουμε το κοινό εγχείρημα, αν έχετε ακόμα κουράγιο. Μη φεύγετε. Μη φεύγετε. Μη φεύγετε. Πάμε να ψηφίσουμε και τα, τα κοινά αυτά εγχειρήματα. Okay, forget about. okay. Καλά, το ξεχνάμε. Yeah. Ja, okay. Also niemand, niemand will mehr, na, es ist wirklich traurig, niemand will mehr... Λυπηρό, λυπηρό. Κανείς δεν θέλει να ψηφίσει άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε αύριο τι ε, ψηφοφορίε ε, με την απαλλαγή τη Κομισιόν 9 η ώρα. 9 η ώρα εννοώ 9. Sorry. I just εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την ψηφοφορία πολύ γρήγορη και σαφής. Το, το καλύτερο κοινό που είχα ποτέ. Λοιπόν, λία τη συνέδρια. Συνεχίζουμε αύριο στις 9 με την απαλλαγή της Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πειθαρχία. Λία τη συνεδρίαση.